για την κατάσταση των κρατουμένων συνέδρια στο Τατζικιστάν. Ε, δίνουμε αμέσως το λόγο στους συντάκτες. Ε, πρώτα η κυρία Χάουταλα. Το Τατζικιστάν είναι η φτωχότερη από τις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας και πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις αυτή τη χώρα. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να υπενθυμίσουμε στη χώρα ότι έχει αναλάβει υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης και Εταιρικής Σχέσης και η συνεργασία μας θα πρέπει να βασίζεται σε κοινέ αξίες. Μόλις χθε από ό,τι γνωρίζω, ο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Τατζικιστάν και Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε χώρα και το Κοινοβούλιο ήθελε να εκπέμψει ένα χειρό μήνυμα ε, για αυτό το διάλογο ήδη μπορούμε να ε, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σημαντική επιδείνωση ε, στην κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε κατασταλτικούς νόμους, ιδίως αυτόν για τις ε, δημόσιες ενώσεις που δημιουργεί σημαντική και ε, απειλές για επιβολή κυρώσεων σε ΜΜΕ. Επίσης, ό,τι αφορά το δικηγορικό σύλλογο, τη δικηγορική πρακτική, υπάρχει ένας νόμος καινούριο που απειλεί την ανεξαρτησία του δικαστικού ε, λειτουργήματος. Και βέβαια έχουμε και το θέμα των πολιτικών κρατουμένων, οι οποίοι καταδικάζονται για φυσικά φανερά πολιτικά ε, κίνητρα πολιτικού λόγου, Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό ούτε και η καταπολέμηση τη τρομοκρατίας πρέπει να δεχθούμε, που βέβαια είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, να μην ε, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταστολή και καταπίεση των δημοκρατικών κόμματων της αντιπολίτευσης. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν το δικαίωμα ε, να υπάρχουν ε, τα φιλιρινικά και δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης και των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Σκοράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είχα την δυνατότητα, την ευκαιρία να παληθεύσω τι συμβαίνει στο Τατζίκισταν, γιατί συμμετείχα στην εκλογική αποστολή που έγινε πέρσι. Και είναι σαφές ότι μιλάμε για μια χώρα με μια πολύ έντονη αυταρχική τάση, όπου οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ή της αντιπολίτευσης δυνατότητα συνέρχεστε και επικρίνει, αλλά και ο έλεγχο του των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι αρκετά σφιχτός. Ε, πλέον έχουμε εταιρική σχέση συνεργασίας με το Τατζίκισταν από το 2009 με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων ε, ε, στόχων, αλλά αυτοί οι στόχοι δεν έχουν διόλου επιτευχθεί. Μάλλον το αντίθετο έχει συμβεί και το συνταγματικό δημοψήφισμα που έγινε πριν από λίγες μέρες, 22 Μαΐου, από, αντικατοπτρίζει στην πράξη ότι ξαλήφονται οι εντολές και ξεπερνάτε το κατόφλι, στρώνοντας το δρόμο για την προεκδική εκλογή του γιου του σημερινού ηγέτη. Και όσον αφορά τους κρατούμενου συνείδηση, θα πρέπει κάπως να υψώσουμε τη φωνή, γιατί έχουμε προνομιακές εμπορικές σχέσεις με αυτή τη χώρα και μπορούμε να επηρεάσουμε. Κύριο Στάνοκ, Πρόεδρε, όπως πολλά με τα κομμουνιστικά κράτη, το Τατζικιστάν έχει περάσει μέσα από μια πολύ επώδυνη διαδικασία αναγέννησης που κόστησε και 100.000 ακόμη ζωές πριν από την δημοκρατική μεταρρύθμιση του 1997. Πολλές από, τις, από τους διχασμούς που βλέπουμε σήμερα είναι ε, υπόλοιπο αυτού του ε, εμφυλίου πολέμου. Ο Ράχμον, ο πρόεδρος, ε, θέλει να επανεκλεγεί για τέταρτη φορά και δεν επιτρέπει τη μετάλλαξη της χώρας προς πιο δημοκρατική χώρα. Συνεργαζόμενος βεβαίως με τη Μόσχα, καταστέλει τη δράση των, ε, της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων, των δικηγόρων. Η εικόνα είναι πολύ ζωφερή. Βλέπουμε το Τατζικιστάν να ξαναπέφτει στο, στην τροχιά ως δορυφόρος της Μόσχας και πολύ περιορισμένες δυνατότητες οι ελπίδες το Ταζικιστάν να στραφεί προς τη Δύση για να εξασφαλίσει τις δημοκρατικές, πολιτικές και οικονομικές προδιαγραφές. Ο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο το Ευρωκοινοβούλιο είχε καταγγείλει το σενάριο στο οποίο είχαν μετατραπεί ε, οι εκλογές ε, για το νέο Κοινοβούλιο του Τατζικιστάν. Ε, Φέτο το Μάρτιο περιοριστήκαν ε, οι εντολέ και επετράπη έτσι στον πρόεδρο Ράχμον που έχει την ίδια θέση από το 1992 να ε, είναι και πάλι υποψήφιο για την Προεδρία. Όχι μόνο είναι δύσκολο το πολιτικό πλαίσιο για να επικρίνει κανεί οτιδήποτε και οποιοδήποτε, επιπλέον έχουν προσθεθεί και ε, δικαστικέ σοβαρέ ε, υποθέσει. Εμεί θα πρέπει να στηρίξουμε την ελευθερία και την ισότητα και προτείνουμε το το θέμα των εμπορικών συμφωνιών που θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχουν όρους, ελευθερία έκφρασης, ε, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι αυτό που, το καθήκον που έχουμε σήμερα σε σχέση με αυτή τη χώρα. Ο κύριος Κέλαμ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, πριν από έξι χρόνια η, ε, συνήφθη η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τατζικιστάν και ε, Έκτοτε έχουμε πολλές οικονομικές ε, σχέσεις. Το άρθρο 2 ωστόσο τονίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και και είναι, αυτές, είναι αυτή που θα πρέπει να διέπει τι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές. Ε, σήμερα υπάρχουν πολύ ανησυχητικά μηνύματα για αυξανόμενη παρενόχληση και καταστολή της ε, αντιπολίτευσης ε, με αποκορύφημα την περασμένη εβδομάδα την καταδίκη δύο μελών τη αντιπολίτευση σε διαβίου κάθυρξη. Συχνά Επίση, παρανοχλούνται οι άνθρωποι που στηρίζουν ε, του όσου κατηγορεί ο κρατικό μηχανισμό και η κρατική εξουσία. Φαίνεται ότι γίνονται και βασανιστήρια. Κατανοούμε τη σημασία των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με τη χώρα αυτή, ωστόσο θα πρέπει όλα αυτά να συνδεθούν περισσότερο με την σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Γι' αυτό και καλό ε, την EIS, την, εξωτερική, την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης, ε, να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να ενημερώνει τους πολιτικούς εταίρους. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάντσες Καλντεντέη το γεγονός ότι υπάρχουν γεωστατηγικά συμφέροντα της Ένωσης σε μια περιοχή, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δικαιολογεί την ανεφόρον στήριξη των ηθινόντων της εν λόγω χώρας, γιατί τελικά αυτό ε, γίνεται κατά δίκη για το λαό, όπως στην περίπτωση του Τατζικιστάν. Με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας η κυβέρνηση καταστήλει την αντιπολίτευση, υπάρχουν ε, αποδείξεις για συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι σχέσεις Ένωσης Τατζικιστάν θα πρέπει να βασίζονται ε, στις γραμμές βιώσιμης ανάπτυξης, ισότητα φύλων, ε, κοινωνία των πολιτών, ενδυνάμωση γυναικών κτλ. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι οι αναδιαναμητικές πολιτικές, η κοινωνική συνοχή είναι σημαντικές πολιτικές για να πάψει ο βίος εξτρεμισμός και κάθε μορφή βίας. Χωρίς δικαιοσύνη δεν θα δοθεί ένα τέλος στη βία. Εμείς έχουμε την ευθύνη να αλλάξουμε το ρόλο που έχουμε στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Γι' αυτό το Τατζικιστάν δεν θα πρέπει να το δούμε απλά σε ένα πιόνι στη σκακέρα. Πρέπει να πάψουμε να κοιτάμε μόνο ε, τα γεωστρατηγικά μας ε, συμφέροντα στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής. Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή. Συνάλφη, κύριε Επίτροπε, η εμβάθυνση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με το Τατζικιστάν είναι πολύ σημαντικό ε, στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον το Τατζικιστάν είναι σημαντικό εταίρο στο πλαίσιο τη στρατηγική ε, για τι σχέσει με την Κεντρική Ασία. Θέλουμε να προωθήσουμε τι επαφέ και τι εμπορικέ μα σχέσει με αυτέ τι ε, χώρε. Είναι και σημαντικό εταίρο το Τατζικιστάν στην καταπολέμηση του φονταμεταλισμού και τη τρομοκρατία. Ε, η χώρα αυτή αναζητεί τη δημοκρατική τη ταυτότητα, βέβαια, 26 χρόνια. Και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται. Οι αρχές ασκούν πιέσει σε ε, ελεύθερα μυαλά, στην ε, αντιπολίτευση, ε, στον τύπο κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, υπάρχουν πολιτικώ υποκινούμενες κατηγορίε, κατά, ε, κατά επικριτών ε, των αρχών και πέραμα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές βρίσκονται στη φυλακή. Θα πρέπει άμεσα να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό το διεθνέ δίκαιο και το δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εγγυηθούν οι αρχέ τη χώρα στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και τώρα παρεμβάσει εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων, εξ ονόματο του ΕΛΚΟ, ο κύριο Στετίνα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι. Το 1992 σταμάτησε ο εμφύλιος πόλεμος στο Τατσικιστάν αφήνοντας πίσω του 30.000 ορφανά. Και το ξέρω πολύ καλά αυτό γιατί στη δεκαετία του 90 προς το τέλος έκανα ένα σχετικό ντοκιμαντέρ ο ίδιος και δούλεψε πάνω σε αυτό. Μεγάλωσαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και θέλησαν να ζήσουν σε μια χώρα όπου θα μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα. Η ελευθερία όμως δεν πνέει στη χώρα αυτή. Οι έννοιες του πλουραλισμού, της δημοκρατίας είναι ξένες στο πολιτικό της πεδίο. Βλέπουμε από τις κατηγορίες και τις ε, ε, φυλακίσεις ε, των πρωταγωνιστών της ε, αντιπολίτευσης Μπουζουρ Μεριόροφ, Νοντήρα Ντοιάνεβα, Νουρεντίν Μαχκάμοφ και άλλων ότι υπάρχουν τόσες παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων Πρέπει λοιπόν ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση ε, στην ε, διάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό πλαίσιο ώστε να βοηθήσουμε αυτούς που διώκονται στο Τατικιστάν. Σοσιαλιστές, Δημοκράτες, Λαουριστίν. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Καλημέρα σας. Όντως, είναι θλιβερό το ότι υποχρεούμεθα να αναγνωρίσουμε πως το Τατζικιστάν είναι ένα από τα κράτη εκείνα του κόσμου που διολυσθένει όλο και περισσότερο προς την αυταρχική διακυβέρνηση το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια λοιπόν ενώπιον του γεγονότος ε, ότι έχει σταματήσει η δημοκρατική ε, αναγέννηση του Τατζικιστάν. Πρέπει να μεριμνήσουμε για ένα δίκαιο σύστημα δικαιοδοτικό και όσο αυτό δεν υπάρχει εκείνοι οι οποίοι ε, θα έπρεπε να προσφέρουν την ε, νομική συνδρομή και υποστήριξη προς τους ε, διοκόμενους, δηλαδή οι συνήγοροι, βρίσκονται οι ίδιοι διοκόμενοι. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το ψήφισμα. Βλέπουμε ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα τις βίες εξτρεμιστικές πράξεις που δεν δικαιολογούνται επουδενή πρέπει να τηρηθούν όλοι οι όροι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποφεύγεται η αδίποτε ε, αυταρχική μέθοδος, η κατασταλτική μέθοδος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ιδιαίτερα να επιμείνει σε αυτά. Ο Πρόεδρος Διακόπτη, ευχαριστώ Γκέρικε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε του Τατζικιστάν. Σήμερα είναι το πρώτο κράτος κεντρικής Ασίας που έχει ε, ανεξαρτητοποιηθεί από τις ε, εταιρικές, εμπορικές σχέσεις, οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, ιδιαίτερα λόγω των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το προγραμματισμό μέχρι το 2020 που καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Τζικιστάν και ακόμη περισσότερο, εάν βέβαια αυτό, ε, αυτό προϋποθέτει να τηρούνται οι όροι και οι συμφωνίες. Γι' αυτό και μας ενοχλεί ιδιαίτερα αυτή η κατάσταση στο και πρέπει να καταγγείλουμε τα προβλήματα όταν η αντιπολίτευση βρίσκεται συλλήβδεν στη φυλακή, όταν η ελευθερία της θρησκείας καταστέλλεται, ε, όλα αυτά είναι ασυμβίβαστα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυρίως, ε, χριστιανικές μειονότητες, οι κυρίως γερμανικές χριστιανικές μειονότητες, σε παραδείγματι, κινδυνεύουν να ε, σβηστεί η, τους, η παρουσία τους στο παρελθόν τους. Ε, πρέπει λοιπόν η συνεργασία με την Ευρώπη να υπάρχει, αλλά να υπάρχει μόνο όταν η δημοκρατία και τα κράτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μια βιώσιμη παρουσία. Στο Τατζικιστάν ο κύριος Σκέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συντάκτες του ψηφίσματος έχουν δώσει μια πολύ καλή περιγραφή για το τι συμβαίνει στο Τατζικιστάν και με το καθεστώς το οποίο ασκείται από τον τωρινό πρόεδρο στη χώρα αυτή. Φυσικά θα πρέπει να συνεργαστούμε με το λαό του Τατζικιστάν αλλά θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση σε αυτούς ώστε να εισαγάγουν μεταρρυθμίσεις και ιδίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της αντιπολίτευσης. Προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και την διαφθορά αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να πριτανεύσουν κανόνες που θα εξασφαλίσουν την ελευθερία του λόγου και η κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές και να ε, ελευθερώσει όλους αυτούς τους κρατούμενους που είναι στη φυλακή. Ο κύριος Φρουντσούλικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι έχουμε κάθε συμφέρον να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ειρήνης και σταθερότητας με την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αλλά οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το Ταζικιστάν συνδέονται με τις κοινέ αξίες για τις πολιτικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό υποστηρίζω απόλυτα την ε, έκκληση για την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων στις φυλακές για πολιτικούς λόγους. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε όταν αυξάνεται ο αριθμό των συλλήψεων και των κρατήσεων και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι εκκρεμούν ποινικά αδικήματα εναντίον τους, αλλά είναι ουσιαστικά πολιτικοί κρατούμενοι. Οι πολιτικοί αυτοί κρατούμενοι, οι δικηγόροι τους, δικηγόροι τους και οι οικοί τους υφίστανται καταστολή. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα μέσα ενημέρωση τα οποία δεν μπορούν να επιτρέψουν την έκφραση ελεύθερης γνώμης, ιδίως για τα σχετικά θέματα. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να εργαστούν ελεύθερα χωρί φόβο κατά δίωξης. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να παρέμβετε για αυτό το θέμα οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό ε, ηγετών της αντιπολίτευσης και υπερασπιστών των δικηγόρων στο Τατζικιστάν. Το ψήφισμά μας επιμένει ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν όλοι αυτοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σε ένα διάλογο, διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Τατζικιστάν και αυτός ο διάλογος θα πρέπει να οδηγήσει και στην εκκίνηση μεταρρυθμίσεων, ιδίω σε ό,τι αφορά ανεξάρτητη δικαιοσύνη με ένα λειτουργικό σύστημα διασταυρωμένων ελέγχων οι δικηγόροι θα πρέπει να μπορούν να εκπροσωπούν ελεύθερα τους πελάτες τους ενώπιον των δικαστηρίων. Και φυσικά πρέπει να έρχονται ενώπιον του δικαστηρίου οι πολίτες του Ταζικιστάν μόνο αν υπάρχουν αξιόπιστες κατηγορίες εναντίον τους και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε διαφανείς διαδικασίες και δίκαια δίκαια. Εγώ χαιρετίζω το έργο του γραφείου του διαμεσολαβητή που παρακολουθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Αλλά παραμένουν πολλά τα οποία χρειάζονται για να υπάρξει απαραίτητη βελτίωση τη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κ. Presidente. Το Τατζικιστάν είναι ένα ιδιαίτερα φτωχό κράτο, όπου όμω υπάρχει συστηματική καταπίεση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών του. Τα μέσα μαζική ενημέρωση, οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών βρίσκονται στο στόχαστο των αρχών επίσης υπάρχει καταπίεση των χριστιανικών πληθυσμών που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα. η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να ασκήσει πίεση στο τατζικιστάν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας του κράτους δικαίου των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης του πολυκομματισμού και της ελευθερίας της έκφρασης. οφείλει η ευρωπαϊκή ένωση να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή στην πράξη του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε και του δικαιώματος σχηματισμού πολιτικών κομμάτων πρέπει επιτέλους να σταματήσει η καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή και νομίζω ότι η ευρωπαϊκή ένωση έχει τα μέσα έχει τον τρόπο και τη δυνατότητα πραγματικά να ασκήσει την πίεσή της προς το τατζικιστάν. ευχαριστώ. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που λόγο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Τατζικιστάν αυτή τη στιγμή είναι η φτώχεια, η πολιτική καταπίεση, ακόμα και βασανιστήρια. Τα μέσα μαζικής ενημέρωση φημώνονται. Ε, πολύ λίγα πράγματα λειτουργούν στη χώρα. Και οι πολίτε δεν είναι ίσοι απέναντι στην κρατική εξουσία. Αυτό δείχνει το πραγματικό πρόσωπο του Τατζικιστάν. Παραδέχομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει με τη χώρα αυτή και η συμφωνία αυτή έχει στατηγική σημασία. Να σας ρωτήσω λοιπόν εάν αυτή η συμφωνία είναι ε, μια κατάφορη άρνηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τελικά. Διότι Το ερώτημα είναι, μπορούμε να εγκαταλείψουμε το, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα λόγω της στρατηγική της σημασίας απλώς. Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς Υποστηρίζω όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ω προαλήσαντε. Εμεί θα πρέπει να υποστηρίξουμε το Τατζικιστάν στον δρόμο τη για την δημοκρατία, ακόμα και αν αυτή η χώρα έχει ένα, επειδή έχει και ένα μακρύ σύνορο με το Αφγανιστάν που παίζει ένα αποσταθεροποιητικό ρόλο. Θέλω να αναφερθώ όμω σε ένα διαδικαστικό θέμα. Αν διαβάσω εγώ το ψήφισμα το οποίο έχω δει, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να στοιχειοθετεί το κατεπήγον. Όλα τα γεγονότα που αναφέρονται είναι εδώ και καιρό γεγονότα. Εγώ με 7 χρόνια στην αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ασίας είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας με το Τατζικιστάν και παρόλα αυτά εγώ δεν είχα καμία ευκαιρία να συμμετάσχω στην εκπόνηση αυτού του ψηφίσματο και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα στο Κοινοβούλιο μα να ξεχωρίζουμε αυτά που είναι πραγματικά ε, επίγοντα και τα θέματα που θα πρέπει να επιληθεί η αρμόδια αντιπροσωπεία ώστε να έχουμε ένα καλύτερο ψήφισμα και να εμπλακούν και άτομα τα οποία γνωρίζουν καλύτερα τη χώρα αυτή. Αν θέλουμε φυσικά οι αντιπροσωπείε του Κοινοβουλίου να έχουν κάποιο νόημα θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτέ τι διαδικασίε. Ο κύριος Καστάλδο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Δυστυχώς το Τατζικιστάν ε, περνάει μια περίοδο που διαπιστώνουμε πολύ συχνά να επισυμβαίνουν στις πρώην Δημοκρατίες. Υπάρχει σχεδόν εμφύλιο πόλεμο. Όχι απλώ αντιπαράθεση μετά του Κομμουνιστικού Κόμματο που έχει την εξουσία και των Ισλαμιστών. Δυστυχώ, σε αυτό το δύσκολο μείγμα απολυταρχία, φτώχεια, ε, λοιπού εσωτερική ασφάλεια και τη απειλή του Αφγανιστάν, το, η ασφάλεια του κράτους βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Αμάλη Ραμών ε, θα ε, έχει αποφασίσει να διώκει τους αντιφρονούντες, ακόμη και τους συνηγόρους ή τους ε, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ως νομικός που έχω λάβει μόρφωση στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα σας έλεγα να μην αφήσουμε να περάσει έτσι η άδικη η δίωξη του Ισλαμικού κόμματος της αντιπολίτευσης είναι έστω και αυτός ένας τρόπος στήριξης της δημοκρατίας. Θα πρέπει να υπάρξει δίκαση και δικαίωμα υπεράσπισης των ανθρώπων αυτών ε, όταν φτάνουν μπροστά στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερο στα πλαίσια της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασία. Οι ρήτρες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να πάψουν να είναι απλά φάσματα και οθόνες ε, ε, καπνού και να γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τηλιανίδη. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε μάρτυρες μιας περίοδου με πάρα πολλές προκλήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για το Τατζικιστάν. Υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις βέβαια τα πρόσφατα χρόνια. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες του συνήγορου του πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρόλα αυτά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά διάφορα ζητήματα. Η κυριότερη ανησυχία μας έχει να κάνει με την πολιτική συμμετοχή και τους πολιτικούς κρατουμένους. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2015 το Ισλαμικό Κόμμα του Τατζικιστάν κρίθηκε εκτός νόμου ως τρομοκρατική οργάνωση και οι επικεφαλής του συνελήφθησαν. Συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητούσε περιορισμό στις δράσεις αυτές. Ζητούμε λοιπόν από την κυβέρνηση του Τατζικιστάν να μην περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως εκείνο της δίκαιας δίκης και να μην ε, διώκει ε, πολιτικά τους ε, πολιτικούς στο Τατζικιστάν. Υπάρχουν ποινές φυλάκισης για 13 ηγέτες του IPT, οι οποίοι έχουν σύλληφθει. Σε δύο περιπτώσεις έχουν καταδικαστεί ισόβια, δυστυχώς. Επίσης, έχουμε εκδώσει δήλωση όπου λέγαμε ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν ήταν αρκετά διαφανής και δεν υπάρχει καμία βεβαιότης ότι πρόκειται για δίκαιες δίκες παρόλο που έχει υπογράψει τις διεθνείς συμβάσεις στο Τατζικιστάν επ' αυτού. Υπενθυμίζουμε επίσης στην κυβέρνηση του Τατζικιστάν ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις αν κατηγορούνται με αδικήματα οι κρατούμενοι. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, Μόνο αν υπάρχει σωστή δικαιοσύνη θα αποφύγουμε τον εξτρεμισμό. Γι' αυτό όλα αυτά τα υπογραμμίζουμε σε πάρα πολλέ συναντήσεις υψηλού επίπεδου που έχουμε. Όταν ο πρόεδρος Ναχμούν είχε έρθει εδώ, στη, πήγε μάλλον στις Βρυξέλλες, και όταν είχαμε και συναντήσεις υπουργικέ ε, πάλι μέσα στο 2015 αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και πολύ πρόσφατα σήμερα μάλιστα επί τη ευκαιρία τη συνάντηση διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ευρωπαϊκή Ένωση στα Τζικιστάν. Τα επαναλάβαμε όλα αυτά. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, η δράση της κυβέρνησης του Τατζικιστάν μπορεί να ζημιώσει την νομιμότητα του πολιτικού συστήματος στο Τατζικιστάν, κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε. Η δικιά μας η πολιτική θέλει να πετύχει πολιτική σταθερότητα και οικονομική ευημερία. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν παραμένουμε κύριος πάροχος αναπτυξιακής βοήθειας τόσο στο Τατζικιστάν αλλά και γενικότερα στην Κεντρική Ασία και θα συνεχίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των κρατούμενων συνειδήσεως να τα βάζουμε πάνω-πάνω στην ημερήσια διαταξή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Τατζικιστάν προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ολοκληρώνεται εκείνη η συζήτηση. Έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφισμάτων. Η ψηφοφορία